Καλησπέρα σας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε μια ωραία αίθουσα με φυσικό φως και επαφή με τον πραγματικό κόσμο. Ας την απολαύσουμε λοιπόν σήμερα. έχουμε στις 4 παρα 10 τις ψηφοφορίες μας. Παρακαλώ μιλισμονέστε τις ε, κάρτες ψηφοφορίας. Και εκτός αυτού το κύριο θέμα είναι η έκθεση του κυρίου Κορέα του Κάμπους για την αμοιβαία συντροπή μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και συνεργασία των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση τη ορθή εφαρμογή των τελωνιακών και γεωργικών μετρητμήσεων. Θα το δούμε αμέσω. Υπενθυμίζω ότι έχουμε ε, μετάδοση της συνεδρίασης από το διαδίκτυο. Καλωσορίζω όλους όσοι μας παρακολουθούν από αυτό. Και επίσης έχουμε ακόμη ένα newsletter του Μαρτίου 2014 της Επιτροπής μας, το οποίο μπορείτε να δείτε. Όποιος δεν το έχει λάβει στο, Συθυρίδα του ή δεν το λαμβάνει, να μας ενημερώσει Όσοι δεν μας παρακολουθούν από το web streaming, επίσης έχουν πρόσβαση από την ιστοσελίδα μας. Θα βρουν άλλωστε όλες τις συνδέσεις για πρόσβαση στα έγγραφα. Υπενθυμίζω στους συναδέλφους ότι έχουμε πρωτοποριακά εισαγάγει την συνεδρίαση χωρίς έγγραφα και μπορείτε να έχετε είτε στον υπολογιστή σας είτε στο τάμπλετ ε, πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και βέβαια σε όλες τις γλώσσες. Πρακτικά, το, οι συνεδρίες 22 και 23 Ιανουαρίου έχουν κατευθεί, θα τα εξετάσετε και αν δεν λάβουμε έως σήμερα το βράδυ σχόλια, θεωρούμε ότι έχουν εγκριθεί. Διαπραγματεύσει τριμερού διαλόγου. Πρόκειται για μόνιμο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Εξέλιξει δεν έχουμε. Η κυρία Σουάλντε Μόζερ που είναι εδώ μας έλεγε την προηγούμενη φορά ότι δεν αναμένεται πρόοδος στο θέμα των σιδηροδρόμων, δυστυχώς. Εμείς ήμασταν από, τον, από τέλειο Οκτωβρίου έτοιμοι να διαπραγματευτούμε το Συμβούλιο. Έχουμε κατά τα άλλα ολοκληρώσει όλα τα κύρια θέματα που είχαμε μέχρι το τέλος της θητείας από την Επιτροπή μας και έτσι μπορώ να προχωρήσω στο μόνο ουσιαστικά εκρεμές νομοθετικό μας θέμα, την πρόταση για κανονισμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για αμοιβαία συνδρομή και συνεργασία όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας σε και γεωργικά θέματα. Έχουμε περίπου 60 τροπολογίες λάβει για την έκθεση αυτή. Και έτσι δίνω το λόγο στον εισηγητή να τη σχολιάσει. Και θα καλέσω στη συνέχεια τους και να να συμβάνουν συζήτηση, όπως και άλλωστε στη συνέχεια μπορεί όποιος άλλος συνάδελφος. Ο κύριος Κοραϊάντε κάπως παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον Πρόεδρο για το 41ο τεύχος του newsletter. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα τεύχη, δεν έχουμε προσωπικότητες, έχουμε ζώα, φυτά και χέρια. Δεν έχουμε φωτογραφίες προσώπων. Οπότε είναι ενδιαφέρον αυτός ο τρόπος, εναλλακτικός τρόπος παρουσίασης των προβλημάτων μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους των πολιτικών ομάδων για το ζωηρό ενδιαφέρον που, έδωσαν, ε, που έδειξαν για την έκθεσή μου. Κάτι που φάνηκε και από το μεγάλο αριθμό των τροπολογιών, 65 το σύνολο. Την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκα με τους ασκιώδης ηγητές για να αναλύσουμε τις τροπολογίες και έτσι μπορέσαμε να ε, συγκλίνουμε τις απόψεις μας και τις περιέλαβα στο έγγραφο της Παρασκευής. Θα το συζητήσουμε και αυτή την εβδομάδα προκειμένου να βρούμε το μέγιστο κοινό παρανομαστή στην Επιτροπή μας ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στις 18 Μαρτίου. Οι τελωνιακοί δεν έχουν μέσα για να ε, διασφαλίσουν κατά πόσο η δηλωμένη προέλευση των ε, ε, προϊόντων ε, είναι η πραγματική και μερικές φορές ε, και τα, ο τρόπος διαμετακόμισης είναι προβληματικός. Φάνηκε ότι έχουμε 1950 περιπτώσεις απατών και άλλων ατασταλιών με αποτέλεσμα να έχουμε γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ ζημίες σε σχέση με την ε, εσφαλή παραπλανητική περιγραφή των ε, ε, μεταφερομένων προβλημάτων Και μάλιστα οι πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος είναι πολύ μεγαλύτερες, γιατί είχαμε πολλές παραβιάσεις, γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι οι ζημίες και έχουμε περίπου 30.000 περιπτώσεις δυνητικής απάτης. Έχουμε δηλαδή ένα παγόβουνο μπροστά μας και εμείς ε, βλέπουμε μόνο την κορυφή. Το υπόλοιπο μάλλον δεν έχει ακόμη ε, ανακαλυφθεί. Και μάλιστα η περίοδος 3, με 7 μηνών για την λήψη των εγγράφων δημιουργεί ακόμη καθυστερήσεις και περισσότερες ζημίες. Και μάλιστα το Ελεκτικό Συνέδριο σε έναν έλεγχο το 2010 ε, λέει ότι με ένα μικρό δείγμα το 200, σε 240 ε, τροπολογίες είχαμε ήδη πολλές, ε, πολλά λάθη και μάλιστα ζημία της τάξης των 58.000 ευρώ. Και μάλιστα α, αυτά τα ποσά δύσκολα ανακτώνται και άρα δεν περιλαμβάνονται στον προπολογισμό της Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες των συναδέλφων, είναι πολύ επικοδομητικές και στόχο έχουν τη βελτίωση της ίουσας νομοθεσίας προκειμένου να γίνει πραγματικός έλεγχος της ε, εισόδου και διαμετακόμισης των εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Ενίσχυονται τα ε, συμφέροντα των καταναλωτών και των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Έχουμε βέβαια και κάποιες προβληματικές τροπολογίες. Έχουμε πολλές τροπολογίες του κυρίου Σβάμπ που ζητά διαγραφή το άρθρο 18 του κανονισμού κάτι που δείχνουν την ανησυχία μας ό,τι αφορά την πρόσβαση στη βάση δεδομένων για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων. Αλλά νομίζω ότι αν ε, επικαλεστούμε την αρχή της προστασίας των δεδομένων, πάση ε, θυσία θα ακυρώσουμε, θα εξουδετερώσουμε το βασικό στόχο της, ε, του κανονισμού. Θα πρέπει απλώς να προσδιορίσουμε τους κανόνες πρόσβασης ε, των κρατών μελών στα διάφορα δεδομένα και της πρόσβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα α, αυτά τα στοιχεία, αντί να διαγράψουμε πλήρως τα άρθρα που ζητά ο κ. από τον κανονισμό. Επαναλαμβάνω λοιπόν, ε, είμαι κατά αυτών των τροπολογιών. Τροπολογίες... Ε, 51 και 84, όλες Σμιτ. Αναφέρουν ένα πρόγραμμα που θα ήθελα να διαλευκάνω. Και πάλι με το επιχείρημα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και του περιορισμού της ε, πιθανής ε, ε, αδικαιολόγητης κυκλοφορίας αυτών των στοιχείων προτείνει εξαντλητικό κατάλογο των διεθνών οργανώσεων στις οποίες θα πρέπει θα μπορούν να λαμβάνονται, να στέλνονται στοιχεία ε, για το περιεχόμενο των εμπορευματοκιβωτίων. Είναι πολύ δύσκολο όμως εκ των προτέρων να προσδιορίσουμε τις διεθνείς οργανώσεις και τους ε, διάφορους οργανισμούς και φορείς ε, που έχουν σχέση με τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και μάλιστα σε συγκεκριμένο χρόνο. Γι' αυτό και το κείμενο αναφέρεται σε ένα μνημόνιο συνεννόηση. Αυτή τη στιγμή ένα οργανισμό ή μια οργάνωση μπορεί να μην έχει καμία σχέση με τα οικονομικά συμφέροντα τη Ένωση, αλλά στο μέλλον μπορεί να έχει τέτοια σχέση, όπω είναι η περίπτωση τη Frontex. Οπότε, χάρη του εν ε, νομοθετήν και προστατεύοντα ταυτόχρονα και τα δεδομένα, δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα εξαντλητικό κλειστό κατάλογο αυτών των οργανώσεων στο κείμενο του κανονισμού είμαι εδώ υπέρ μιας μεγαλύτερης ελαστικότητας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη βάση για τις ε, συμβαστικές λύσεις ε, που εξέτασα με τους σκιώδεις ηγητές την περασμένη Παρασκευή και που θα συζητήσουμε αυτή την εβδομάδα, αποτελείται αυτή η βάση από εννέα συμβαστικές τροπολογίες που προσπαθούν να διασκεδάσουν τις ανησυχίες των συναδέλφων σε ένα συνεκτικό και χρήσιμο κείμενο που θα εξυπηρετεί τους στόχους μας και που τους προανέφερα. Δηλαδή την προστασία των καταναλωτών, που είναι και τελικοί αποδέκτες ε, αυτών των προϊόντων που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ταυτόχρονα και προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η δύο στόχη που θέλω να καλύψω με τις τροπολογίες. Οι συμβαστικές τροπολογίες που αφορούν το άρθρο 18H και που μιλάει για τις ε, προϋποθέσεις από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί άμεσα να ζητήσει από τους οικονομικούς φορείς ε, τις πληροφορίες, βρίσκονται σε αρχική φάση. Στόχος ε, είναι να επιστρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να μπορεί να το κάνει σε περίπτωση που κολλησιεργούν τα κράτη-μέλη. Είπαμε ότι τρεις εβδομάδες δίνονται στα κράτη-μέλη για να αποφανθεί και να ικανοποιήσει το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν μιλήσουμε για σιωπηρή παραπομπή, δηλαδή να μπορεί να στραφεί άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους οικονομικούς φορείς. Βέβαια θα πρέπει να επεξεργαστούμε περαιτέρω το κείμενο για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το στόχο μας και να γίνεται σωστή χρήση της βάσης των δεδομένων. Πάντως πιστεύω ότι είμαστε σε θέση να, να πούμε ότι είμαστε αισιόδοξοι ότι θα φέρουμε σε αίσιο πέρα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Πιστεύω ότι η συνετική λύση στην οποία θα, θα πρέπει να καταλήξουμε θα πρέπει να είναι σφαιρική και μόνο τότε θα είναι έγκυρη Κάτι που προϋποθέτει υποχωρήσεις από όλα τα μέλη και μέρη. Γι' αυτό ε, θα ήθελα να ζητήσω από όλους να δείξουν συνεργάσιμο και διαλεκτικό πνεύμα. Μάλιστα η ομάδα μου είναι πρόθυμη να αποσύρει το τμήμα που αφορά τις εισαγωγές από το πακέτο αυτό προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα ηχηρό μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο στην Ολομέλεια του Απριλίου, τότε που θα ψηφίσουμε την έκθεση. Οπότε θα μιλούμε για εισαγωγές και διαμετακόμιση εμπορευμάτων και αν συμφωνήσουμε θα, θα αποκλείσουμε τις εξαγωγές. Αυτό είμαστε διαδεθειμένοι να κάνουμε, να αφαιρέσουμε τις εξαγωγές και να περιοριστούμε μόνο στις εισαγωγές και τη διαμετακόμιση. Αύριο στις ε, 10.30 έχω προγραμματίσει συνάντηση με τους κοιοδησηγητές και ευελπιστώ ότι θα έχουμε σημαντική πρόοδο στις συζητήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε, ας ακούσουμε τους σκιώδεις εισηγητές. Ο κύριος Ροτ ε, πρώτος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την δουλειά που έχει κάνει. Νομίζω πως πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ακόμα δεν έχω δει τα σχέδια συμβαστικών τοπολογιών προτείνεται. Ελπίζω να καταλήξουμε γρήγορα σε κάποιους συμβιβασμούς. Οι βασικές μου παρατηρήσεις. Όσον αφορά την δυνατότητα της Κομισιόν να λαμβάνει αμέσως πληροφορίες από εταιρείες. Άρθρο 18 AIDS. Είναι κάτι το ευαίσθητο γιατί εμείς θέλουμε να προστατεύουμε και τους πελάτες ε, και τις εταιρείες. Οι συνταστικές τροπολογίες 7 και 8 νομίζω είναι επαρκής λύσης. Εγώ θα προσέθω τα δύο πραγματάκια τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Ε, στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών. Κατά την άποψή μου τώρα οι διαβουλεύσεις μεταξύ κομισιών και εκπροσώπων του κλάδου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων νομίζω πως είναι ένας καλός τρόπος για να αναπτύξουμε κάποιες ε, πράξεις ερώτηση στο άρθρο 18F. Δεν ξέρω αν σκοπεύετε να βάλετε τις διαβουλεύσεις αυτές στις συμβαστικές σας τροπολογίες. Τέλος θα ήθελα να επιμείνω στις ε, διευκρινήσεις που έχω βάλει ε, στην τροπολογία 42 και στα σχετικά έγγραφα για το τι είναι παραστατικό στην τροπολογία 43 επί του άρθρου 12. Νομίζω πως πρέπει να γίνει σαφές αυτό για να μην έχουμε κάποια σύγχυση. Ευχαριστώ να τα συζητήσω αυτά με τον κύριο τεκάμπος και τους άλλους συναδέλφου της επόμενης εβδομάδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Ρος. Ο κύριος Σμιτ νομίζω απουσιάζει, δεν ήρθε μάλιστα. Κυρία Ριούλε. Θα είμαι σύντομη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον εισηγητή για τις συμβαστικές προτάσεις. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τις υποστηρίζουμε. Κύριε Ashley Fox. Ο σχεδοσηγητής για την ομάδα μας μου έχει δώσει μια δήλωση και υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία ήθελε να σας ευστήσω την προσοχή και προφανώς σας στείλω αντίγραφο στον εισηγητή. Έχει να πει λοιπόν τα εξή. Ε, ήταν ικανοποιημένο με το επίπεδο συνεργασίας και τη της αρχής συμφωνεί με τους στόχους της πρότασης ε, της Κομισιόν, έχοντας όμως δει το ζήτημα πάρα πέρα και λαμβανωμένων των δεδομένων θεωρεί πως οι προκλήσεις είναι αξεπέραστες και ε, λέει τα εξή για να το τεκμηριώσει αυτό. Πρώτα απ' όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη δημιουργία ενός κεντρικού αρχείου για τα ζητήματα αυτά πηγαίνουν πάρα πολύ πιο πέρα από αυτό το οποίο καθορίζει η Κομισιόν στην μελέτη αντικτύπου και το βασικό είναι πώς θα επιβάλλουν τα κράτη-μέλη την μεταφορά αυτών των δεδομένων εάν αρνηθούν οι εταιρείε ή εάν στείλουν ανεπαρκή στοιχεία. Δεύτερον, επισημαίνει πως δεν θα μπορέσει να αποδεχτεί την πρόταση για άμεση πρόσβαση από την Κομισιόν στις εταιρείε. Έχει καταθέσει κάποιες τροπολογίες στο άρθρο 18H ε, και αυτές τι θεωρεί το ελάχιστο που θα μπορούσε να δεχτεί, αλλά θα προτιμούσε την τροπολογία του κυρίου Σβάμπ επί του 18C, γιατί η διαγραφή αυτού του άρθρου κατ' ουσίαν ε, διαγράφει την ιδέα περί ενός τέτοιου μητρώου. Και νομίζω και ο Σβάμπ θεωρεί πως αυτό καλύπτεται από άλλα δεδομένα νομίζω από τη μεταρρύθμιση του τελωνιακού προγράμματος. Μετά συνεχίζει ο κύριος Φόξ. Η αξιολόγηση της Κομισιόν Λάθος υποθέτει πως δεν θα υπάρχει κόστος ε, εφαρμογής από τα κράτη-μέλη για την παροχή αυτών των δεδομένων. Η... Ο συντονισμός των διαφόρων συστημάτων πληροφορικής των κρατών μελών είναι κάτι το οποίο θα κοστίσει και δεν είναι δυνατόν να γίνει μια σωστή ανάλυση χωρίς να ληφθεί υπόψη αυτό το κόστος. Όσον αφορά τις τροπολογίες, θεωρεί πως οι τροπολογίες ε, που αφορούν την ε, καταγέρα και θάλασσα μεταφορά δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν γιατί βεβαίως το σύστημα έχει δημιουργηθεί έχοντας κατά νου τις χερσαίες μεταφορές οπότε το να επεκταθεί σε άλλου τύπου μεταφορές ε, είναι κάτι το οποίο απαιτεί πρώτα απ' όλα μία διαβούλευση. Επίσης το 18α ε, η διαχείριση κινδύνου σημαίνει και τυχαίους ε, δειγματοληπτικούς κινδύνους. Ε, επίσης αναφέρεται σε δραστηριότητες όπως κατανομή πόρων που είναι εθνικές αρμοδιότητες και η διαχείριση κινδύνου εδώ πέρα θα δημιουργήσει σύγχυση για τον ρόλο της Κομισιόν και των κρατών μελών. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως ο κύριος Φόξ ανησυχεί πως η Κομισιόν δεν έχει σκεφτεί επαρκώς ε, τις επιχειρησιακές ε, προκλήσεις και θεωρεί πως χρειάζεται πιο λεπτομερής εξέταση εάν είναι να ξεπεράσει αυτά ο τελικός κανονισμός. Αυτή είναι η πρόταση του κυρίου Φόξ. Τώρα, ποιος άλλος θέλει να μιλήσει, ο κύριος Σβάμπ. Έχετε καταθέσει πολλές τροπολογίες, η κυρία Λεγκρίπ, όχι, η κυρία Γκέπχαρτ και ο κύριος Σβάμπ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ ιδιαίτερα στον εισηγητή για την ε, τοποθέτησή του τελευταία στιγμή στην ε, τροπολογία μου την προηγούμενη εβδομάδα. Βλέπω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε την συνεργασία στο πνεύμα που έχει προεξαγγείλει. Και εδώ με τις τροπολογίες του βλέπουμε ότι μπορούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ ιδιαίτερα στο άρθρο 18 και να πω ότι δεν αμφισβητεί κανείς από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι σε τέτοιου είδου ρυθμίσεις, κανονισμούς έχουμε να κάνουμε πάνω απ' όλα με το ποιος θα έχει προσβάσει σε ποιες πληροφορίες. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει, θα πρέπει να έχει ένα νέο πεδίο πρόσβασης, δυνατότητες πρόσβασης εδώ και το σύστημα και την προηγούμενη εβδομάδα με το e-call, είπαμε ότι θα πρέπει να ρυθμίσουμε και τα θέματα των λοιπών ενδιαφερομένων και δικαιούχων με κάποιο τρόπο λογικό, ρεαλιστικό και γι' αυτό θα έλεγα ότι δεν θα πρέπει να έχουμε μια βάση δεδομένων στην οποία να μπορεί η Επιτροπή ανα πάσα στιγμή της διαδικασίας απεριόριστα να έχει πρόσβαση σε δεδομένα ακόμα και δεδομένα που δεν έχουν καμία σχέση με τις θελωνιακές υπηρεσίες. Και γι' αυτό συμφωνούμε με τον κύριο Κορείαντε Κάμπος να αναζητήσουμε μια λύση η οποία να αφορά ακριβώς εκείνες τις πληροφορίες τις οποίες, στις οποίες θα μπορεί να έχει πρόσβαση η Επιτροπή αλλά να τις προσδιορίζει με πιο σαφή τρόπο. Εάν πούμε δηλαδή ότι θέλουμε να έχουμε περισσότερες δυνατότητες για πρόσβαση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατανοεί και τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται στα θελωνιακά θέματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ καλά, αλλά να μην τη δώσουμε και εν λευκό επιταγή. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο λογική λύση. Πολύ ευχαριστώ λοιπόν να συνεργαστώ με τον εισηγητή κύριε Πρόεδρε, ώστε να βρούμε την καταλληλότερη διατύπωση. Πάντως ευχαριστώ πολύ που δεν απέρριψε απλά και μόνο την τροπολογία μου, αλλά προσπάθησε να βρει μια λύση. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ την όλη υπόθεση αν μπορέσουμε και στην προσεχή θητήρα να συζητήσουμε πώς θα το χειριστούμε το θέμα και ελπίζοντας ότι θα έχουν τα κράτη-μέλη και τη διάθεση να ε, προσεγγίσουν προς τώρα τις θέσεις μας όπως και σε άλλα σημεία. Ευχαριστώ πολύ και θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια συγκεκριμένη λύση λοιπόν για διατύπωση. Ευχαριστώ κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ Πρόεδρα. Ευχαριστώ τον Αντώνιο Κορέα Πολύ καλή η δουλειά. Και για να κάνω μια προκαταβολική παρατήρηση. Δεν κάναμε απλώ μια παρεμπίπτουσα παρατήρηση, κύριε Σφαπ. Μιλήσαμε με πολύ ξεκάθαρου όρου ε, για την προστασία των δεδομένων. Το ποια δεδομένα μπορούν να μεταφέρονται και σε ποιο βαθμό είναι δυνατόν να διαβάζονται προσωπικά στοιχεία των ατόμων που επιβαίνουν στο αυτοκίνητο. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήθελα να καταστήσω απόλυτα σαφές πριν αρχίσουν να διαδίδονται μέσω του διαδικτύου εσφαλμένες πληροφορίες. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι συμπληρωματικά. Βλέπω ότι πολλές τροπολογίες προβλέπουν τη διαγραφή ε, διατάξεων που έχουν να κάνουν με την προστασία των δεδομένων. Με επιχείρημα ότι ούτως ή άλλως η οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ισχύει δεσμευτικά και άρα δεν χρειάζεται να γίνει επιπλέον αναφορά της. Πολύ καλά. Και έστω. Ερωτώ όμω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε θέση να μας εξηγήσει γιατί έχει διατυπώσει αυτές ε, τις ζητάξεις κατά αυτόν τον τρόπο. Ήταν πράγματι η καταλληλότερη επιλογή να μπει μέσα στο διατακτικό του κειμένου ή μήπως ίσως στο, στις αιτιολογικές σκέψεις να ήταν σκόπιμο να κάνω μια παραπομπή στην οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Έχω ιδιαίτερη ε, ανησυχία να μην κάνουμε τίποτε λάθος στην υπόθεση αυτή για τα προσωπικά δεδομένα. Ο Πρόεδρος, θέλετε να λάβετε το λόγο κάποιος άλλος συνάδελφος πριν δώσετε το λόγο στην Επιτροπή. Και βέβαια μετά και στον εισηγητή. Όμως πρώτα θα ήθελα να καλωσορίσω μια ομάδα επισκεπτών της κυρίας Σάλντε Μόζερς, μια ε, συναδέλφου που δουλεύει πολύ σκληρά και αποτελεσματικά στην Επιτροπή μας, σοσιαλδημοκράτες από την Νότια Δανία, εκεί στα αριστερά και τους χαιρετούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και συγχαρητήρια και χειροκροτήματα. Very good. Λαμπρά. Ο κύριος Γιαννάκης, αν δεν κάνω λάθος, από την Όλαφ που είναι επιφορτισμένος με το δοσιά αυτό, θα μας κάνει κάποια σχόλια. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με κάλυψαν οι προελίσσαντες τα περισσότερα και ήδη διαφαίνονται κάποιες συμβαστικές λύσεις και μάλιστα έχουν συνταχθεί και όλα μερικές. Εγώ θα επικεντρωθώ στα μείζωνα κατά τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέματα. Έχουμε καταρχήν τις ε, τροπολογίες 55-56 και επόμενες που αναφέρεται στα CSMs και τις τροπολογίες 79 και τις υπόλοιπες που μιλάνε για εισαγωγές, εξαγωγές και διαμετακόμιση. Κατά τη γνώμη μας είναι απαραίτητο να έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα μέσα να ανοιχνεύει και να βοηθήσει καλύτερα τη δίωξη σε περίπτωση απατών που αφορούν εισαγωγές, εξαγωγές και διαμετακόμιση. Και για το λόγο αυτό χρειάζονται τα CSM, στα, τις πληροφορίες αυτές για τα εμπορευματοκιβώτια και τα στοιχεία για εισαγωγές και εξαγωγές, καθώς και για διαμετακόμιση. Το κόστος για τις, για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με την παροχή αυτών των στοιχείων θα είναι ελάχιστο, γιατί ήδη έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτό που λέμε global dump, δηλαδή να στείλουν τα πάντα από τους υπολογιστές τους ε, με ένα απλό κλικ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε είναι τελείως ε, ε, ανευκόστος αυτή η διαδικασία της παροχής των στοιχείων. Επίσης, ήδη γίνεται κάτι τέτοιο ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι τελωνιακές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών λαμβάνουν από τους μεταφορείς προειδοποιήσεις για όλες τις εξαγωγές ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι εισαγωγές ε, προς τις Ηνωμένε Πολιτείες ε, είναι γνωστές και μάλιστα 48 ώρες πριν την άφηξή τους στην Αμερικανική επικράτεια από τα στοιχεία που δίνουν οι μεταφορείς στις τελωνιακές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή ήδη έχουν τέτοια εμπειρία οι μεταφορείς. Μπορούν αντίστοιχες πληροφορίες να τις διαβιβάζουν και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε τελική ανάλυση και στα κράτη-μέλη σε όποιον άλλο φορέα τις χρειάζεται γιατί είχαμε επαφές ε, με εκπροσώπους της, ε, εκπροσώπους ε, των μεταφορέων και πιστεύουμε ότι τέτοια διαβίβαση πληροφοριών μπορεί να γίνει χωρίς κόστος για τις επιχειρήσεις. Επίσης αποδείξαμε και στο παρελθόν ότι είναι πολύ, σημαντική, πολύ σημαντικά τα στοιχεία διαμετακόμισης και εισαγωγών ίσως ε, δεν είναι τόσο γνωστή η χρησιμότητα και τις βάσεις δεδομένων για τις εξαγωγές και για τα στοιχεία εμπορευματοκιβωτίων που εξάγονται. Και αυτό το θέμα οδήγησε ακριβώς στην πρόταση, στην ιδέα ότι ίσως ε, δεν είναι απαραίτητα τέτοια στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή δηλώσεις εξαγωγών ή CSM εξαγωγών. Εγώ θα σας εξηγήσω τώρα γιατί απαιτούμε και, γιατί ζητούμε και αυτά τα στοιχεία των εξαγωγών και εσείς θα σταθμίσετε κατά πόσο είναι χρήσιμα αυτά τα δεδομένα και πόσο σημαντικά είναι ή αν υπερέχει η χρησιμότητα αυτών των δεδομένων από την πιθανότητα κατάχρησης κάποιων δεδομένων. Είναι δύο είδη τα είδη των απατών. Σε πολλές περιπτώσεις είδαμε ότι οι εισαγωγές γίνονται μόνο και μόνο με πρόθεση την επανεξαγωγή αλλά παρόλα αυτά τα αγαθά παραμένουν σε ευρωπαϊκή επικράτεια. Κάτι που σημαίνει ότι ο Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και κυρίω ο προϋπολογισμός των κρατών μελών χάνει έσοδα από ειδικού φόρου κατανάλωση και από φόρο προστιθέμενης αξία. Αυτό είναι το ένα είδο απάτης. Δεύτερο είδο απάτης είναι όταν αγαθά υποτίθεται ότι θα, θα εξαχθούν, αλλά στην ουσία επανέρχονται ω αντικείμενα λαθρεμπορίου. Δεν είναι σπάνιο αυτό το φαινόμενο. Πρόσφατα είχαμε μια, ένα ανακοινωθέν τύπου για σημαντική κατάσχεση από τις Ισπανικές αρχές μεγάλου φορτίου σιγαρέτων που υποτίθεται ότι είχαν εξαχθεί από την Κύπρο ε, με προορισμό τη Βολιβία και στο μεταξύ έμειναν λαθρέα επέστρεψαν λαθρέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι ότου τα ανακάλυψαν οι Ισπανικές αρχές και τα κατάσχεσαν. Τέτοιου είδους λοιπόν απάτες μπορούν να ανοιχθούν πολύ πιο εύκολα εφόσον έχουμε στην διάθεσή μας και δηλώσει εξαγωγών και στοιχεία για τα εμπορευματοκιβώτια, τα CSM εξαγωγών. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι απαραίτητα και τα στοιχεία για τις εξαγωγές. Βέβαια, εσείς θα σταθμίσετε τη σχέση χρησιμότητας και κινδύνων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την άμεση πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε έγγραφα, κυρίως τιμολόγια και άμεση επαφή με τους οικονομικούς φορείς. Αυτό που ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να έχει τα έγγραφα. Δεν θέλουμε κατά ανάγκη να στρεφόμαστε άμεσα στους οικονομικούς φορείς. Μπορούν να μας τα δίνουν και τα κράτη-μέλη. Τα έγγραφα μας ενδιαφέρουν. Οπότε μια αναδιατυπωμένη πρόταση ε, για το 18H, αν μπορεί να ε, επιτύχει αυτό το στόχο, δεν έχουμε καμία αντίρρηση με την αναδιατύπωση. Θα ήθελα πάντως να επισημάνω ιδιαίτερα στην τροπολογία 95 που στο τέταρτο εδάφιο αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να στραφεί άμεσα στους ε, ιδιώτες, ε, στους ιδιωτικούς ε, οικονομικούς φορείς, εκτός για τα κράτη-μέλη αρνούνται την παροχή του εγγράφου. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό, γιατί μπορεί με η τροπολογία να δεν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να αναδιατυπωθεί για να αποφευθεί η διακριτική ευχαίρεια στα κράτη-μέλη είτε να απορρίψουν την ε, αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε να την αναβάλουν, να αναβάλουν την ικανοποίηση της επαόριστον. Αυτά και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα στον εισηγητή γιατί οι προτάσεις με την τελευταία τους διατύπωση προσθέτουν ε, ρεαλισμό και επαναφέρουν μια ισορροπία στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτικότατη απάντησή σας. Τώρα, αν δεν θέλει κάποιος άλλος να παρέμβει, γιατί έχουμε λίγο χρόνο, θα ζητήσω από τον εισηγητή να απαντήσει σε αυτά τα οποία είπατε και σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακούστηκαν για να δούμε τι θα γίνει με τις συμβιβαστικές ε, τροπολογίες. Οπότε, κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τους και οδησυγητές και τους υπόλοιπους συναδέλφους και πάνω απ' όλα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δική της παρέμβαση. Συνήθως, όταν επεξεργαζόμαστε ένα κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσπαθούμε να συγκλίνουμε τις απόψεις, γιατί μπορεί αρχικά να υπήρχε μεγάλη διάσταση απόψεων, αλλά στην πορεία των συζητήσεων ερχόμαστε όλο και πιο κοντά και μειώνεται αυτό το χάσμα. Τώρα έχουμε μια περίεργη κατάσταση. Σε μερικές περιπτώσεις είχαμε τέτοια προσέγγιση και τέτοια σύγκληση. Και μερικέ τροπολογίε επιτρέπουν αυτή τη σύγκληση των απόψεων, όπω με τι τροπολογίε του κυρίου, με τροπολογίες του κυρίου Σβά. Πιστεύω ότι εκεί θα καταλήξουμε σε συμφωνία και σε μείωση των διαφορών. Σε άλλε περιπτώσει όμω φαίνεται ότι διευρύνεται αυτή η διάσταση των απόψεων, απομακρυνόμαστε ακόμη και από την αρχική πρόταση και από τι αρχικέ μα συζητήσει με τους κοιόδε ηγητέ και οι τροπολογίες των μεταρρυθμιστών και συντηρητικών είναι σήμερα πολύ πιο απαιτητικέ και πιο ακραίες από τις αρχικές. Απ' την άλλη πλευρά θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι εν μέρη το επιχείρημα της προστασίας των δεδομένων δεν ευσταθεί γιατί εδώ δεν μιλούμε για προσωπικά δεδομένα, δεν μιλούμε για δεδομένα που έχουν σχέση με πρόσωπα, αλλά με κινήσεις εμπορευμάτων. Και είναι 4-5 δείκτες ουσιαστικά που μιλούν για την προέλευση του εμπορευματοκιβωτίου, το περιεχόμενό του, διαμετακόμιση, ημερομηνία Αποστολή, ημερομηνία άφηξη, Αυτά είναι τα στοιχεία. Δεν έχουν σχέση με πρόσωπα, με προσωπικά δεδομένα. Γιατί λοιπόν επικαλείστε την ιδιωτική σφαίρα ή την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Είναι ψευδοδήλημα αυτό. Ούτως ή άλλως στην Αλία η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν συνάπτει συμφωνία με μια χώρα, με τη Χιλή για παράδειγμα, κάθε αλλιευτικό σκάφος που αλλιεύει στα χωρικά ήττα της Χιλής οφείλει να δηλώσει τα CSM για να έχει δικαίωμα εκφόρτωσης ε, του αλλιεύματος. Και έτσι έχει πρόσβαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτά τα CSM. Οπότε είναι... πληροφορίες έχουν υλικό περιεχόμενο. Δεν σχετίζονται με πρόσωπα ή με προσωπική ζωή. Μπορεί κάποιες πληροφορίες να έχουν στρατηγικό ενδιαφέρον για κάποιες πληροφορίες και να είναι πρόθυμα τα κράτη-μέλη να κυκλοφορούν. Για παράδειγμα, οικονομικές πληροφορίες για την αξία των εξαγωγών. Αυτό το καταλαβαίνουμε, ότι τα κράτη-μέλη μπορεί να είναι επιφυλακτικά ή τουλάχιστον μερικά κράτη-μέλη είναι επιφυλακτικά απέναντι στην διακίνηση τέτοιων πληροφοριών. Αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε Έχουμε ούτω ή άλλω πάρα πολλέ εισαγωγέ και εξαγωγέ, εσόδου και εξόδου. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μερικέ από αυτέ ε, να διαταράσουν, να παραβιάζουν την κοινοτική νομοθεσία και να στοιχειοθετούν ε, απάτε. Άλλωστε, παραλαμβάνω, πρόκειται για διακινήσεις ε, εμπορευμάτων και δεν επιτείνεται με την πρόταση αυτή η γραφειοκρατία γιατί η μεταφορά των δεδομένων γίνεται απλώς με ένα πάτημα κουμπιού, με ένα κλικ. Εμείς, επαναλαμβάνω, χάρη διαλλακτικότητας και ανέβρεση συμβαστική λύση θα μπορούσαμε να θυσιάσουμε τις εξαγωγές παρόλο που συμφωνούμε ότι χάνονται τις σημαντικές πληροφορίες αλλά αυτό το κάνουμε μόνο χάρη συμβασμού και σύγκλησης. Βέβαια θα πρέπει να αναγνωρίσω ότι χάσαμε πολλές ώρες στην κοινοβουλευτική θητεία, αφιερώσαμε πολλές ώρες στη συζήτηση του προπολογισμού της Ένωσης για την επόμενη επταετία και δεν είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε ότι ε, η, τα έσοδα από τους θελωνιακούς δασμούς που είναι από τους ελάχιστους ίδιους πόρους που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνονται ε, έρμεο των απατών. Γιατί ούτως ή άλλως Ξέρουμε ότι υπάρχουν απάτες, ξέρουμε ποιε είναι οι ζημίε και απώλειες για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, έχουμε μηχανισμούς να τις αποτρέψουμε και αντί να το κάνουμε επικαλούμαστε κάποια ψευδοδιλήμματα ή κάποιες ανύπαρκτες απειλέ. Κύριε Πρόεδρε, μερικές προτάσεις μπορεί να ανοίγουν το φάσμα των ευκαιριών και των δυνατοτήτων. Αλλά μερικές άλλες, όπως το κύριο Σφάμπ, επιδέχονται κάποιων μικρών βελτιώσεων και αναδιατύπωση προκειμένου να ληφθούν υπόψη. Εγώ δεν είμαι απεσιόδοξο, θεωρώ ότι είμαι ρεαλιστή και πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε στη συμφωνία και ευελπιστώ ότι θα διαπεράσουμε αυτό το θέμα κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, κοιτάξτε, όπως ξέρετε πρέπει 18 Μαρτίου να ψηφίσουμε γιατί τότε είναι η τελευταία μας ευκαιρία να εγκρίνουμε κείμενο για να προλάβουμε την δεύτερη ολομέλεια του Απριλίου. Ε, νομίζω έχουμε ήδη βρει μια θέση για την έκθεση Υπάρχουν λοιπόν σχεδόν 15 μέρες που φτάνουν ε, για τις διαπραγματεύσεις. Είμαι σίγουρος πως θα μπορέσουμε να, να τα καταφέρουμε και θα μπορέσει μετά και το Συμβούλιο να τα δει. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν. Κοιτάξτε, ε, είμαστε και πέντε λεπτά νωρίτερα από την ώρα μας, αλλά μια που ψηφίζουμε θα κάνουμε ένα διαλυματάκι, οπότε μη φύγετε. Μέχρι να μαζευτούν όλοι οι βουλευτές για την ψηφοφορία. Θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε ακριβώ παρά 10. Και βέβαια χρειάζεται και τις κάρτες σας για να ψηφίσετε. Ευχαριστώ πολύ τον Σίτη. Uh, to take your places, uh, Παρακαλώ καθίστε για την ψηφοφορία. Θα ήθελα να καλωσορίσω κάποιους ε, καλεσμένους που βρίσκονται στην ψηφοφορία. Ε, δεν είναι και πολύ συναρπαστικό, αλλά εν πάση περιπτώσει σας καλωσορίζω στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Τώρα έχουμε δύο θέματα για τα οποία δεν έχουν κατατεθεί τροπολογίες για τις ε, τελωνιακές ε, παραβιάσεις και κυρώσεις θα ήθελα να ζητήσω από τους ηγητές να πούν δύο λόγια αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να ψηφίσουμε για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων του τριμερού διαλόγου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υποπίεση. Ήταν πολύ έντονος ο τριμερής διάλογος γιατί κάποια κράτη-μέλη θεωρούσαν πως ήμασταν κατά των βασικών σημείων της ε, ενιαίας αγοράς αλλά τελικά συμφώνησαν με την θέση μας. Ε, κύριε Σφάμπ, κατάλαβα καλά, εσείς θα κάνετε την παρουσίαση ή εγώ. Εσείς. Καλώς. Κοιτάξτε, ήμουν πρόεδρος στον τριμερή διάλογο. Καταλήξαμε σε μια αρκετά καλή συμφωνία. Δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Έπρεπε να επανέλθουμε τελικά και να σας υπενθυμίσω πως όπως με όλα αυτά τα πακέτα νομοθεσίες αναδιατύπωσης το Κοινοβούλιο ήθελε να διαφυλάξει τα συμφέροντά του ειδικά όσον αφορά την ε, πρόσβασή μας στις ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων παράλληλα με τις ε, διαδικασίες ε, πράξεων κατεξιοδότηση. Και οπωσδήποτε θα θυμάστε πως η Κομισιόν είχε κάποιες αντιρρήσεις στην διατύπωση, κατά έχουν κάνει για πολλωστή φορά, εν πάση περιπτώσει είναι ένα ζήτημα που θα αντιμετωπίσει το επόμενο κοινοβούλιο. Λοιπόν, αν δεν θέλει κάποιο άλλο να πει κάτι, τίθεται σε ψηφοφορία ηλεκτρονική νομίζω, έτσι. Έρχεται η κάρτα του κυρίου Σουάμπ, θα τον μετρήσουμε, εν πάση περιπτώσει. Σας παρακαλώ λοιπόν να υπερψηφίσετε την θέση μας στον τριμερή διάλογο, έρχεται η ψηφοφορία. 29 κάρτες υπάρχουν, αλλά 28 μόνο ψηφίζουν. Κάποιος δεν πατάει το κουμπάκι. Πέρας. 27 υπέρ. Ε, μία αποχή, μία ψήφος κατά. Οπότε θα πάει νομίζω στην Ολομέλεια τη δεύτερη του Απριλίου. Ωραία. Περνάμε τώρα σε ένα σημαντικό σχέδιο ψηφίσματος για μια νέα πρόταση που λάβαμε από την Κομισιόν για τις τελωνιακές παραβάσεις και σχετικές κυρώσεις. Οι συντονιστές αποφάσισαν πως δεν υπάρχει χρόνος για μια πλήρη έκθεση, αλλά είναι αρκετά σημαντικό το θέμα για να κάνει κάποιες πολιτικές δηλώσεις η Επιτροπή, οπότε εμπιστευτήκαμε τον εισηγητή μας για το θέμα αυτό, την κυρία Λιγκρίπ δηλαδή και την κυρία Γκέπχαρτ που επίσης παρακολουθούσε το θέμα ως και εισηγήτρια. Είναι λοιπόν διακομματική η άποψη και συμφώνησαν και οι άλλες πολιτικές ομάδες. Αλλά αν θέλετε μπορείτε να κάνετε μια σύντομη εισαγωγή. Ξεκινάμε από την κυρία Λεγκρίπ. Oui, merci, monsieur. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο λόγια πολύ γρήγορα πριν να περάσουμε στην ψηφοφορία για, την, για το ψήφισμα αυτό για ένα κοινό ψήφισμα για τις κυρώσεις, τις τελωνιακές κυρώσεις και παραβάσεις. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Γκέπχαρτ για το πολύ καλό κλίμα συνεργασίας καταρχάς, το οποίο μπορέσαμε να αναπτύξουμε. Κατά τη διατύπωση αλλά και τη διαπραγμάτευση του σχέδιου ψηφίσματος, σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεννόησης για το κοινό καλό με το ΣΥΠΗΝ εργαστήκαμε. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα, αλλά και τους κοιόδης ηγητές που μας έδωσαν τις παρατηρήσεις τους και τις τροπολογίες. Προσπαθήσαμε να τις ενσωματώσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό στο τελικό κείμενο. Ελπίζω ότι επετεύχθη ο στόχος και ότι θα έχουμε την ευρύτερη δυνατή υποστήριξη για το ψήφισμα. Στο ψήφισμα αυτό θέλω να υπενθυμίσω ότι δεν επισήλθαμε σε όλες τις ε, νομικές αλλά και πρακτικές λεπτομέρειες που αφορά ε, που αναφέρει η πρόταση για το νομικό πλαίσιο της Επιτροπής, γιατί θέλουμε να παραδώσουμε τη σκητάλη στην προσεχή θητεία, στην προσεχή σύνθεση της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ. Απευθύνουμε έκκληση δηλαδή και παραδίδουμε τη σκητάλη. Ώστε η προσεχή ΣΥΜΚΟ να αναλάβει το καθήκον να εξετάσει με μεγάλη προσοχή την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επιθυμία μας είναι η σημερινή ψηφοφορία να προχωρήσει κατά τρόπο συνεπή και με την ε, τελευταία μεταρρύθμιση του τελωνιακού κώδικα και να επαναλάβει για άλλη μια φορά τη βούλησή μας για μια πραγματική τελωνιακή ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που αποτελεί για μας έναν πυλώνα για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ την κυρία Λογκρίπ, τη συνάδελφο, για την πολύ καλή συνεργασία των ομάδων μας ε, και βέβαια τη γραμματεία. Στο ψήφισμα αυτό έχουμε καταγράψει ταχύτητες ρεκόρ και εξεύρει συνενέσεις όπως συμβαίνει καμιά φορά όταν ε, συνεργάζονται διαφορετικές ε, πολιτικές ομάδες, δεν θεωρείται αυτονόητη η συνένεση και η συμφωνία. Αλλά εδώ τα καταφέραμε. Όπως είπε η κυρία Λεγκρίπ, εδώ διατυπώνουμε πολιτική κατεύθυνση χωρίς όμως να υψερχόμεθα σε λεπτομέρειες. Και έτσι τροπολογίες από τις διάφορες ομάδες οι οποίες υψερχόνταν υπερβολικά στις ε, λεπτομέρειες δεν ε, έγιναν δεκτές και επειδή υπάρχουν διαφορετικές ε, θέσεις, νομική βάση και το καθεξής. Και γι' αυτό είπαμε ότι στα διαφιλονικούμενα ζητήματα δεν παρεμβαίνουμε, κοιτάμε μόνο τι χρειάζεται να εμβαθύνουμε με το ψήφισμα αυτό και αφήνουμε για το επόμενο κοινοβούλιο το καθήκον της εξέτασης των λεπτομεριών για να είναι συνεπέζευε το αποτέλεσμα και καλό. Με το κείμενο αυτό σήμερα πιστεύω έχουμε σήμερα μια καλή και σαφή θέση για καλύτερη και σαφέστερη συνεργασία στον χώρο των τελωνίων και εκφράζουμε ταυτόχρονα θέσεις για το θέμα των κυρώσεων και γενικά τη συνεπούς αντιμετώπιση αντίστοιχων περιπτώσεων. Αυτά είναι τα ζητήματα που είχαμε. Και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία και στην προσεχή να δούμε μπροστά μας και πάλι το κείμενο αυτό, να το επεξεργαστούμε για να ετοιμάσουμε ένα καλό νομοθέτημα και να συνεχίσουμε έτσι αυτή την πολύ σημαντική δουλειά. Ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά που έχετε κάνει. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσει η Επιτροπή την θέση της. Τίθεται λοιπόν σε ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία ε, επί του σχεδίου ψηφίσματος. 30 συνάδελφοι ψηφίζουν. Αν μπορείτε λίγο γρήγορα. Σβάμπ, ναι. Πέρας. 29 Πέρα. Ε, μία ψήφος κατά, σαφές ζητήσαμε να ψηφιστεί στην, ολομέλεια, στην πρώτη Ολομέλεια του Απριλίου και να σας πω, κυρίες Γκέπχαρτ και Λεγκρίπ, φροντίστε να το μάθουν οι γραμματείες των πολιτικών ομάδων σας γιατί θα πρέπει η διάσκεψη των πρόεδρων να μας δώσει χρόνο συζήτησης και αγόρευσης. Πρέπει λοιπόν να είναι και ο Επίτροπος παρόν και οπωσδήποτε ένας ομιλητής από την κάθε πολιτική ομάδα. Α, μπορώ να το υπογράψω λοιπόν τώρα και θα πάει και στους εισηγητές και μετά στις υπηρεσίες της Ολομέλειας. Η Έλενα θα σας το φέρει και ο κύριος West πέρα από την Κομισιόν είναι εδώ, οπότε διαπιβάστε κι εσείς το ότι θα θέλαμε να έρθετε να κάνετε μια παρουσίαση και να αντιδράσετε κάποια στιγμή. Ωραία. Περνάμε τώρα στις πιο ουσιαστικές ψηφοφορίες ε, στην έκθεση διασπορβουλίας για την προστασία των ε, καταναλωτών στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Θέλετε να πείτε κάτι κύριε Βάριν Χόλτσερ, όχι. Ωραία. Περνάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. it's kind of you to since I'm the Oh no, Emma is here, but. Um... Ναι, ναι, είναι η εδώ. Ε, μια που ψηφίζω και εγώ και είμαι σκιώδης ηγητής, ε, πρέπει να φροντίσω να ψηφίσω σωστά. Ε, ευχαριστώ λοιπόν για την υπομονή σας. Λοιπόν, συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Οπότε περνάμε στην τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 30 υπέρ κατά απορρίπτεται 31, 32, 33 υπέρ κατά δεκτή αλλά να τις επαληθεύσουμε γιατί είναι σημαντικές να δούμε αν λειτουργούν και τα συστήματα Άρχεται η ψηφοφορία για τις 31, 32, 33 γίνονται δεκτές. Ωραία. 37 καταπίπτει, οι επόμενες δύο επίσης. 36 καταπίπτει. 38 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 39. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 45 υπέρ. Κατά δεκτή. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά δεκτή. 48 υπέρ, κατά δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά δεκτή. 52 υπέρ, κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 7. Με προφορική τροπολογία. Εντάξει, δεν έχετε πρόβλημα, ωραία. Συμβαστική 7 με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε στην 61 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 63 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 64 υπέρ κατά απορρίπτεται 65 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβιβαστική 8 υπέρ κατά δεκτή 74 υπέρ κατά δεκτή 75 υπέρ κατά απορρίπτεται 76 υπέρ κατά απορρίπτεται 77 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβαστική 9 υπέρ κατά δεκτή και περνάμε στις 84 και 85 ταυτόσιμες υπέρ κατά δεκτή δεκτές 86-87 κατά καταπίπτουν. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 91 με την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 92 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 94 και 95. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 96 αποσύρεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 101-102 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 103-104 καταπίπτων. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τροπολογία 110 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τροπολογία 115 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 116 υπέρ. Κατά δεκτή. 118-117 καταπίπτων. Συμβιβαστική 14 υπέρ. Κατά δεκτή. 124 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 15 σε δύο μέρη, όπως ζήτησε η Άλντε. 15 μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Δεκτό. Μέρος δεύτερο. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά να είμαστε σίγουροι. Ναι. Εδώ αν είστε και ξύπνοι κιόλας. Απορρίπτεται το δεύτερο μέρος. Οπότε περνάμε στην 132 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβιβαστική 16 υπέρ κατά δεκτή 137 υπέρ κατά δεκτή 138 και 139 υπέρ κατά δεκτή 140 και 141 να ψηφίσουμε 141 ως προσθήκη. Α, προσθήκη στην 140. Μάλιστα. Οπότε περνάμε στην 142. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 143 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά. Δεκτή.

κυρία Στάιλερ ως προσθήκη υπέρ. Όχι. Όχι, 154 έγινε δεκτή. Οπότε μπορεί να γίνει ως προσθήκη σε αυτή. Όχι. Καταπίπτει. Ωραία. 156 λοιπόν υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 1 έχει αποσυρθεί περνάμε στην εκτελεστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 3 υπέρ κατά δεκτή τροπολογία 4 υπέρ κατά δεκτή στις αιτιολογικές σκέψεις ε, τροπολογία 5 υπέρ κατά Δεκτή. 6 και 7 κατά καταπίπτουν. 8 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά δεκτή. Το 21 υπέρ. Κατά επίσης δεκτή. 22 πίπτη Οπότε ψηφίζουμε τώρα για αυτό για την έκθεση πρωτοβουλίας. έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή με 27 υπέρ, μία ψήφο κατά, δύο τροπολογίε. δύο αποχές βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και νομίζω πως θα πάει στην ε, Ολομέλεια. Στην τελευταία Ολομέλεια αυτής της θητείας, πότε θα είναι η τελευταία έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας αυτής της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Τελειώσαμε για σήμερα. Η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 17 και 18 Μαρτίου. Να σας υπενθυμίσω, στις 17 Μαρτίου έχουμε την ακρόαση για το TTIP, την συμφωνία, στις 3 η ώρα και έχουμε εξαιρετικούς ομιλητές μεταξύ των οποίων και επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρώπης και τον ΙΠΑ που θα έρθουν και οι δύο. Οπότε πραγματικά δεν πρέπει να το χάσετε θα μεταδοθεί στο διαδίκτυο. Σας περιμένω λοιπόν στις 17 Μαρτίου 3 η ώρα και βεβαίως θα έχουμε και το επόμενο απόγευμα συνέχεια στις 3 η ώρα. Θα τα λάβετε σε ένα email. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα.